Bueno, uh, querida... Αγαπητοί συνάδελφοι, για να δούμε όσοι δεν έχουν την πρόθεση να κάνουν επεξηγής ψήφου, ας ακενώσουν ε, την αίθουσα. Τώρα, αν θέλουν να κάνουν ε, σώνει και καλά ιδιωτικές συνομιλίες και πηγαδάκια πριν το γεύμα, Εντάξει, εμείς θα περάσουμε σε επεξηγήσεις ψήφου πάντως, που είναι πολύ άριθμες. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον Ντανιέλ Χάναν, που θα μας εξηγήσει την ψήφα του για την έκθεση της κυρίας Γκυγιόμ για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Κύριε Χάναν, έχετε το λόγο.